Καλώ welcome colleagues. Sorry I'm a few minutes late. Uh, hope you Καλώς ήρθατε συνάδελφοι. Συγγνώμη που καθυστέρησαμε λίγο. Ελπίζω να μην το βάλατε ήδη στο Twitter ότι άργησε η Πρόεδρος. Εντάξει, δεν ήταν ε, υπονοούμενο. Μπορείτε να το βάλετε αν θέλετε. Συνήθως ε, είμαι εδώ πρώτη, αλλά δεν τα κατάφερα. Θεωρώ ότι υιοθετείται η ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ωραία, ευχαριστώ. Ε, έγκριση των πρακτικών της 14ης ε, Οκτωβρίου 2013 συγγνώμη, εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στο σημείο 3, έκθεση του Jean-Paul για ε, την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία. Να του δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με όλη αυτή την κοσμοσυρωή ε, σήμερα στην αίθουσα και τον αριθμό των δημοσιογράφων φαίνεται ότι το θέμα που εξετάζουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικό για την, διάταξη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ουσιαστικά έχει ως στόχο να επιφέρει τροποποιήσεις στον κανονισμό για ε, την ε, κοπή νομισμάτων ε, ε, δεν είναι θέμα ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή των Εθνικών Τραπεζών. Ουσιαστικά μιλάμε για το πάχο των νομισμάτων, των κερμάτων και τη αναδιατύπωση που απαιτείται. Το Κοινοβούλιο δίνει τη γνωμοδότησή του για το πάχος ε, των κερμάτων γιατί ήδη η διάμετρος και το βάρος τους ε, έχει ε, ήδη επιληθεί ως θέμα. Ουσιαστικά λοιπόν επικεντρωνόμαστε στο πάχος. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να αναφέρω. Θα ήταν μόνο ενδιαφέρον να συμπεριλάβουμε στις ιδεολογικές σκέψεις ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την αποφυγή της παραχάραξης και να, αν υπάρχουν ε, περαιτέρω τροποποιήσεις να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Έκανα κάποιες ε, τροπολογίες όμως ξέρω ότι στις ε, προηγούμενες περιπτώσεις που έχει εξετάσει το Κοινοβούλιο καμία τροπολογία δεν έγινε δεκτή. Σταματώ εδώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε ο Ζαν Μπεσέ θα μου στείλει μου έστειλε κάποιες ε, απολογίες επειδή δεν βρισκόταν εδώ σήμερα, ε, γιατί είπατε δεν πρόκειται για θεμελιώδες ζήτημα για την Ευρώπη. Εγώ βεβαίως δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είπε κιόλα ότι δεν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημείο καμπή ε, για την ευρωπαϊκή ιστορία. Ενώ θεωρώ ότι η απουσία του αποτελεί σημείο καμπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Οι σκιώδει δεν παρευρίσκονται. Κάποιος άλλος. Σβέν, έχει το λόγο. Ζήτησα να αντικαταστήσω τον Ζαν Πολ που ήδη έτυχε τόσο θερμής υποδοχής από τους ε, συμπατριώτες του. Όμως ε, Στηρίζουμε πλήρως τις τροπολογίες και συγχαίρουμε τον Ζαν ε, γιατί σε, αυτές τις, ε, σε αυτή την έκθεση είχε ακόμα και την πρόθεση να επιφέρει αλλαγές. Συγχαρητήρια λοιπόν Ζαν Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Λοιπόν, φαίνεται ότι έγινε η εξέταση του σχεδίου. 14 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της 5 Δεκεμβρίου και θέλουμε να ψηφιστεί την ίδια ημέρα και να πάει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Ζωάν Πολ, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Όχι. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, όπου όμως ε, δεν είναι εδώ οι αρμόδιοι. Τι υποτίθεται ότι θα συζητούσαμε μισή ώρα το θέμα των, ε, των κερμάτων. για να μιλήσουμε τόση ώρα για αυτό το θέμα, θα έπρεπε να βάλουμε κέρματα, όπως τα jukebox. Συγγνώμη, συνάδελφοι, φαίνεται ότι έχουμε κερδίσει περίπου 30 λεπτά. Να περιμένουμε τουλάχιστον να έρθει εδώ ο εισηγητής. Ο Σάιντα Αλκαντρεουή και σε ισχυώδεις εισηγητές από τις υπόλοιπες ε, πολιτικές ομάδες. Έχουμε μισή ώρα λοιπόν. Okay, we've waited until the appointed... Ωραία. Περιμέναμε μέχρι που να φτάσει η ώρα που είχαμε ορίσει εκ των προτέρων πριν να φτάσουμε στις προτάσεις για τις κοινοτοπιστωτικές αγορές. Ο εισηγητής μας είναι εδώ, ο Σαΐντ Εντσάιντ, Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, πρόταση κανονισμού για τα εμβέα κεφάλαια της χρηματαγοράς. Ο εισηγητής είναι ο Σαΐντ Αλκαρντούι. Θα σας δώσω το λόγο για να προβούμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε και έχετε δίκιο, πρόκειται για την πρώτη εξέταση γενική συζήτηση για αυτόν τον κανονισμό που προτάθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την... Ε, ε, α, συγγνώμη, διακόπτη Πρόεδρος. Λαμβάνω μια γλώσσα που δεν είναι τα αγγλικά στο κανάλι 2. Ελπίζω τώρα να δουλεύει η ερμηνεία. Ωραία. Στις 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ε, κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συγγνώμη, ενέκρινε ε, μια δέσμη με την ανακοίνωση για την προσέγγιση του σκιώδους τραπεζικού κλάδου και μια συγκεκριμένο κανονισμό για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Η διαχείριση αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων αφορά χίλια δισεκατομμύρια ευρώ, επομένω πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα του τραπεζικού κλάδου και σε φορά και τη βαρχιπρόθεσμη ε, χρηματοδότηση και επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και κρατών. Από οικονομική σκοπιά λοιπόν ε, είναι εξαιρετικά χρήσιμος κλάδος και θέλουμε πλέον αυτόν τον κλάδο να τον ρυθμίσουμε πιο συγκεκριμένα. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα, στις επόμενες εβδομάδες ε, το σχέδιο ε, έκθεσής μου θα οριστικοποιηθεί και θα εξεταστεί στις 2 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ε, για την κατάθεση τροπολογιών. Έχει τεθεί προθεσμία για τις 10 Δεκεμβρίου και στις 20 Ιανουαρίου θα τα εξετάσουμε και η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή και τον Απρίλιο θα έχουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σε αυτούς τους δύο μήνες θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να δούμε και με το Συμβούλιο αν ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για να οριστικοποιηθεί ε, το, ο φάκελος αυτός πριν από το τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης. Βεβαίως έχουμε την κρίση των χρηματαγορών, και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς ε, υπήρξαν θύμα αυτή τη ε, κρίση Με την επτώση της Lehman Brothers ε, κατακριμνίστηκαν και αυτά. Και ξέρετε ότι σε μερικές μέρες 300 δισεκατομμύρια δολάρια βγήκαν από την αγορά και αυτό αφορούσε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες χρηματαγορές, ε, πολλά κράτη-μέλη δέχτηκαν σημαντικές πιέσεις με σημαντικούς ε, συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα αμοιβά κεφάλαια, αλλά και με τον κλασικό τραπεζικό κράδο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς ε, θα ελαχιστοποιήσουμε ή και θα απαλείψουμε αυτούς τους συστημικούς κινδύνους. Μπορεί να θυμάστε ενδεχομένω ότι το 2010, πριν από το ΕΣΜΑ, ξεκινήσαμε με, την, ε, με τον ακριβή ορισμό αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων και εκεί υπήρξε διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και ε, κανονικών, αν θέλετε, τέτοιων αμοιβαίων κεφαλαίων και δόθηκε ορισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Προς το παρόν ε, διεξάγονται σημαντικές συζητήσεις και με τους σκιώδεις. Ελπίζω να λάβω και σημαντικές πληροφορίες από τους σκιώδεις. Όμως πολλά από τα σημεία τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα την χάνουν στήριξή μα και συνάγουν και με τη θέση ε, που υιοθετήσαμε πέρυσι στην έκθεση για τον σκιώδη τραπεζικό κλάδο στο σύνολό του. Και εκεί αναγνωρίσαμε και τον σημαντικό ρόλο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ιδιαίτερος όμως αναφερθήκαμε ε, στα, στα σύννευς, αυτά που έχουν εγγενή αξία και που κάποιες φορές ε, είναι ευάλωτα. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τα ενισχύσουμε και να καλύψουμε τον κίνδυνο και το ρίσκο ε, ρευστότητας. να περιορίσουμε τους κινδύνους που συνδέονται με, τον, με τους εγγενείς κινδύνους και να ε, εντάξουμε και να σωματώσουμε και το κόστος και να έχουμε αυτή την εγγενή αξία με άλλες μεθόδους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτή τη πτυχή. Και αυτό ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, απαγορεύει, δεν μας εμποδίζει αυτά τα σύναυς να τους ε, ενσωματώσουμε και μια τέτοια εγγενή αξία που μπορεί ε, να περιορίσει τις μεταβολές, να τα μεταφέρουμε λοιπόν όλα αυτά σε ε, μεταβλητά κεφάλαια, όμως θεωρεί ότι αυτά τα σύναυς για να περιοριστεί ο κίνδυνος φυγής θα πρέπει να έχουν ένα buffer, ένα παθηματικό ασφάλειας, τουλάχιστον 3% του ε, περιοσιακού στοιχείου. Αυτή είναι η λύση που προτείνει η Κομισιόν. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η απαλληφθεί αυτόν τον ε, σύναυς και να μην επιτρέπεται σε κανένα αμοιβαίο κεφάλαιο να ε, περνάει στην μεταβλητή φάση στη μεταβλητή μορφή αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων για να αποφεύγονται και οι μεταβολές και διακυμάνσεις για τους επενδυτές. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τραπεζική άδεια, bank license, και εκεί βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος ε, όρων και προποθέσεων που θα πρέπει να καλύπτουν οι τράπεζες. Μετά, ο κλάδος ε, εξετάζει αυτό το liquidity fee, όμως βλέπουμε ότι αυτό μετακυλείται στους επενδυτές και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, σε περιπτώσεις ε, κρίση, όταν οι επενδυτές θέλουν να διαρρεύσουν, θα πρέπει να καταβάλουν ένα τέλος. Όμως και πάλι αυτό δεν αποτελεί λύση γιατί θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο κίνδυνος ε, μαζικής φυγής. καλό τους ε, συναδέλφους βάσει της πρότασης της Επιτροπής ε, να εργαστούμε περαιτέρω και να δούμε αν αυτή η ιδέα του αποθεματικού ασφαλείας, του buffer, μας δίνει επαρκείς εγγυήσεις ή εάν πρέπει να κινηθούμε περαιτέρω ε, στην ε, υποχρεωτική μεταβολή. Αυτό θα εξεταστεί στις επόμενες εβδομάδες. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο σίγουρα θα ανακύψει είναι ο ρόλος των ratings. Αρχικά η πρόταση της Κομισιόν ήταν ότι τα σύναυς ιδιαίτερα να μην ζητούν ε, τέτοιο rating και ο συλλογισμό τη Επιτροπή είναι ότι τα σύναυς δεν θα πρέπει ε, να αξιολογούνται γιατί στην πράξη μόνο ε, ε, τριπλό α μπορούν να πάρουν ως αξιολόγηση γιατί σε άλλη περίπτωση αυτό θα προκαλέσει απευθείας μαζική φυγή με τις συναφείς ζημίες. Μια άλλη πτυχή, το ζήτημα της αξιολόγησης είναι η πρόταση της Επιτροπής να μην δίνουμε, δείχνουμε και μεγάλη εμπιστοσύνη στους οίκους αξιολόγησης, αλλά να ενισχύσουμε την δική μας ε, ικανότητα αξιολόγησης ε, των προϊόντων ε, και των τραπεζών. Και προβλέπεται μια ολοκληρή διαδικασία για αυτό το σκοπό. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικό σημείο συζήτησης αυτό το θέμα της εσωτερικής αξιολόγησης. Ουσιαστικά θεωρούμε ότι μέσα από αυτά τα ποιοτικά μέτρα που προτείνονται, δηλαδή διαφοροποίηση επενδύσεων, ε, οι κανόνες ρευστότητας, οι κανόνες ε, ε, συγκέντρωσης, περιορισμοί και αυτό το αποθεματικό κεφαλαίου, όλα αυτά τα μέτρα μαζί λοιπόν, ουσιαστικά θα πρέπει να οδηγήσουν στην αποφυγή των κινδύνων ή μεγάλων κινδύνων φυγής. Ακόμα τρία σχόλια ίσον σημασίας. Όλα αυτά συνδέονται και με τη διαφάνεια βεβαίως. Πολλά στοιχεία του κανονισμού είναι καινούργια και θεωρούμε ότι αυτό είναι θετικό. Θα μπορούσαμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε, για παράδειγμα, για αυτόν τον ρόλο ε, αξιολόγησης και τον τρόπο ε, υπολογισμού αυτών των τελών, μετά ε, το ζήτημα της εποπτείας, του φορέα εποπτείας, στο πλαίσιο της, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας θεωρήσαμε ότι θα πρέπει οι μεγάλες τράπεζες να τεθούν υπό εποπτείες. Αυτό θα πρέπει να γίνει και για τα μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια. Γιατί πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται δεκάδες ε, δισεκατομμύρια ευρώ και ίσως έπρεπε να ε, τα επιτηρούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, σίγουρα θα πρέπει να γίνει και η διασύνδεση με τους χορηγούς και τον κλασικό τραπεζικό κλάδο. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό πώς ακριβώς, ε, ποια είναι η επιρροή των αμοιβαίων κεφαλαίων στον κλασικό τραπεζικό κλάδο στο παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο για να μην ούτως ώστε οι ε, μεταβολές ε, ή ε, αναταραχές στα αμοιβά κεφάλαια να μην επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τον παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο. Αυτά ήθελα να πω εν συντομία. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί καλή βάση για μένα καλή βάση συζητήσεων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα, μια συνολική συμφωνία πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Αυτό θα ήταν θεσπέσιο για να έχουμε στον οδόν το συντομότερο και την κατάλληλη εφαρμογή αυτών των μέτρων. Και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους για να καταλήξουμε σε μια καλή και εξισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Σα uh, uh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Από πλευρά Λάμπερτ ζητήθηκε να μπορούσε να παρέμβει γιατί έχει πάει. Μπορούμε να δώσουμε τον λόγο Ζαν Πολ στον Φιλίπ. Είναι λοιπόν γενναιόδος ο Ζαν Πολ. Φιλίπ, επιτρέπεται λοιπόν τώρα να μπορείς να παρέμβεις εσύ, παρακαλώ. Προφανώς ε, θα πας κάπου και έχεις αυτή την υποχρέωση. Λοιπόν, οι δυνάμεις του κακού δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στις θέσεις και στα σημεία όπου αναμένεται να βρίσκονται. Τουλάχιστον δεν είναι πάντα εκεί. Ας ξαναβρω τις σημειώσεις μου πάλι, για να μην πω καμιά νοησία. Μια στιγμή παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι άγορες ε, σε σχέση με αυτά τα ιδρύματα είναι σχεδόν τραπεζικά ιδρύματα ιδιαίτερα όσον αφορά τα money market funds. Και γι' αυτό η παραδοσιακή οδός είναι ότι αν κάνει κανείς κάτι τότε εκτίθεται στους ιδίους κανόνες αν κάποιος εκτίθεται στους ιδίους ε, κινδύνους πρέπει να καλύπτεται με τους ίδιους κανόνες και κανονισμούς ώστε σε σχέση με τα όσα ο Επίτροπος Μπαρνιέ τη σοφία του αποφάσισε να πράξει ότι Απεφάσισε δηλαδή ότι ουσιαστικά θα εκτίθενται σε 3% όσον αφορά το κεφαλαιακό αυτό, τον κεφαλαιακό αποσβεστήρα και θα πρέπει στο CRD4 να εντάσσονται σε σχέση με κανόνες και κανονισμούς ή θα ε, εντάσσονται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις ε, σε σχέση με το 3% όσον αφορά την μόχλευση το ποσοστό μόχλευσης. Ένα σημαντικό πράγμα που δεν είδαμε στην πρόταση της Επιτροπής και θα έπρεπε πιστεύουμε να εντάσσεται είναι η αντικυκλική πτυχή στις απαιτήσει ε, για αυτές ε, τις ε, διατάξεις. Έχουμε δει ότι είναι πολύ ευμετάβλητα τα πράγματα όσον αφορά τις αλλαγές των αγορών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το να εντάσσονται λοιπόν σε ένα συνετό πλαίσιο αντικυκλικών αντιμετώπισης ε, των, ε, της κυκλικής ε, επαναφοράς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα και θα πρέπει φυσικά να εξετάσουμε και να δούμε αν θα έχουμε κάποιες προθεσμίες μια και βλέπουμε ότι είναι σαν τα τραπεζικά ιδρύματα να δούμε αν θα πρέπει να εντάσσονται σε εξειδικευμένες άδειες με κανόνες και κανονισμούς, μεταφράζοντας δηλαδή αυτές τις ειδικέ απαιτήσει με τέτοιου είδους αδειοδότηση. Κάνουμε λόγο και για τις μεταβατικές περιόδους. Πρέπει να είναι το δυνατόν συντομότερες και να ευθυγραμμίζονται με το CAD 4 αυτές οι διατάξεις. Επίσης θα θέλαμε να περιορίσουμε την ενδυνάμει έκθεση όσον αφορά τα παράγωγα, για παράδειγμα, γνωρίζοντας ότι Βασικά γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ο πιο ευμετάβλητος τομέας των παραγόγων και δεν θέλουμε να αυξηθεί ο συστημικός κίνδυνος που ενέχει εδώ. Τι άλλο να προσθέσω? Μάλιστα. Κάπως ε, μας ε, εκπλήσει το γεγονός ότι η αρμόδια εποπτική αρχή Ευρωπαϊκή Αρχή ΣΕΣΜΑ και πάλι βλέποντας τα EMF έχουμε πολύ συναφείς κατασκευές όπως τα τραπεζο, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες. Σκεπτόμαστε μήπως η EBA δεν θα έπρεπε να εξετάζει, να καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να υπάρχουν διαφορετικοί διαφορετικές παραδόσεις εποπτείας ε, και θέλουμε να είναι τα πράγματα σε ένα ενιαίο συναφές πλαίσιο. Οι προτάσεις μας θα αντανακλώνται στις τροπολογίες ώστε να υπάρχει διαφάνεια για την καλύτερη εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτών των ιδρυμάτων. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Αυτά θα μεταφραστούν το δυνατόν ταχύτερα σε τροπολογίες και θα υπάρξει το δυνατόν να έχουμε, η δυνατότητα να έχουμε το, την μεγαλύτερη διάδραση, αμφίδρομη δράση σε σχέση με τον εισηγητή, ώστε να μπορέσει και να επιταχυνθεί, να προαχθεί η διαδικασία. Και πάλι ευχαριστώ, Ζαμπόρ, που μου επέτρεψες να παρέμβω πιο πριν. Salut. Right, thank you. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σιλβί. Α, χάνω το μυαλό μου. Ο Ζαν Πόλ είναι ο πρώτος που πρέπει να μιλήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το μοναδικό πρόβλημα του να απαρίσταται κανείς πάντοτε είναι ότι δεν τον βλέπουν. Όταν είναι κανείς μία διαρκής παρουσία το ξεχνάνε. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, για να ενθαρρύνω τον εισηγητή στην αποφασιστικότητα που επέδειξε, Δεν θέλω να του πω ότι συμμερίζουμε απόλυτα την αισιοδοξία του για το χρονοδιάγραμμα. Πραγματικά θα ήταν καλό να μπορέσουμε να τελειώσουμε πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Θα πρέπει βεβαίως να τονίσουμε ορισμένα σημεία. Υπάρχει το πρόβλημα του ποσοστού του ε, κεφαλαιακού αποσφεστήρα, καθώς και άλλα θέματα. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι με λίγο όταν ακούω την Επιτροπή να προτείνει την απαγόρευση του να ζητηθούν αυτονομίσματα. Ξέρετε ότι ήμουν εισηγητής των δύο πρώτων ε, εισηγήσεων ο ε, συγητής συνάδελφο Ντομινίκη ε, ε, Μπίτσι και νομίζω ότι υπάρχει μία αντίφαση μεταξύ του να μην θέλουμε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχουμε εντάξει αυτό το επάγγελμα εξασφαλίζοντας μία εποπτεία σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να μας απασχολήσει αυτό το θέμα, γιατί αν το κείμενο ε, μπορεί να προβλέψει ότι δεν μπορεί να ζητηθούν ακατονομίσματα, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει να υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να διακρίνει κανείς με έναν αστερίσκο, για παράδειγμα, τα πλαστά υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εκδίδουν καρτονομίσματα ή κάνουν αξιολογήσεις και τι να μην επιτρέψουμε σε αυτούς που τώρα είναι οργανωμένοι για να μπορούν να παρέχουν καρτονομίσματα ποιότητας. Αυτά είναι τα σημεία που με απασχολούν και πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Σε Ό,τι αφορά τα υπόλοιπα δεν θα έφτανα μέχρι το σημείο που έφτασε ο Φίλιπ Λάμπερκ που θα επιθυμούσε να γίνει το Ταμείο Τράπεζα και να εφαρμοστεί ο κανονισμός των τραπεζών. Ε, δεν θα έλεγα να περάσουμε σε ένα σύστημα χωρίς ρύθμιση, σε ένα σύστημα με υπερβολική ρύθμιση. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι με χαροποιεί πάρα πολύ αυτή η έκθεση με τον, του εισηγητή με τον οποίο έχω ιδιαίτερα καρποφόρες επαφές. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Σιλβή. Ευχαριστώ Σαρα, θα μιλήσω γερμανικά. Α, η πρόταση είναι να συνεχίσουμε το διάλογο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ντοσχέ. Θα ήθελα να πω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτυγχάνουμε τον στόχο του Απριλίου ή χανόμαστε στην μετάφραση. Ο κύριο Κλίμ συνυπέρ των προσπαθειών που γίνονται από την Επιτροπή. Πιστεύω ότι το σημείο αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Θα επιθυμούσε να προσέξουμε ιδιαίτερα το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Πιστεύει ότι Είχανόμαστε θα πρέπει να είναι του κυριου κλιμ συνυπερ προσπαθειων που γινονται απο την επιτροπη πιστευω οτι το σημειο στόχος αυτής της επένδυσης. Ξεγνωρίζει ότι οι έχουν ε, αποδίδουν μεγάλη σημασία στην προσβασιμότητα έχουν ε, οι επιπτώσεις είναι συγκεκριμένες όταν υπάρχουν κυκλικές ίση αγοράς θα πρέπει το MMF δεν ε, αρνήθηκε να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα επενδυτών λαμβάνοντας ε, υπόψη ορισμένα στοιχεία θα πρέπει ε, να παρέχεται επιπλέον κακιολική ρευστότητα για να καλύπτεται το πλαίσιο και θα πρέπει να πούμε ότι οι διατάξεις των και των θα πρέπει να θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν και θα πρέπει να υπάρξουν και ε, ορισμένες ε, προβλέψεις από πλευράς εποπτικής αρχής. Πιστεύω ότι η σύντομη συζήτηση που έχουμε μας δείχνει ότι τα μηδέ κεφάλαια, τα, τα μη αυτά δεν είναι τράπεζες βεβαίως, από τη μία πλευρά θα ήταν γελίο να αυξήσουμε τα απαιτούμενα, τις απαιτήσει ε, για κεφάλαια και να αφήσουμε ανοιχτέ αυτέ τι τράπεζε. Από την άλλη πλευρά δεν δημιουργούμε μία δεύτερη κατηγορία τραπεζών. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, εξετάζαμε την έκθεση Μακάρθη, Υπήρχαν τρεις αρχές επί των οποίων συμφωνήσαμε. Η πρώτη ήταν να σταματήσει αυτή η διάσωση, τη δεύτερη να ε, έχουμε τη βεβαιότητα να είναι αξιόπιστες οι οδηγίες και μετά να, υπάρχει, να υπάρχουν ορισμένα λογιστικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, για μία ακόμα φορά δεν καταφέρνουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύο, τα, αυτά τα βασικά ε, προβλήματα που προσπαθούμε να ε, επιλύσουμε υπήρξε μια επικάλυψη στον τομέα το λογιστικό εκεί που οι τράπεζες είναι χορηγοί και όπως είπε η Σίλβη θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ των τραπεζών και των, ε, Πέρα από ότι δεν αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα υπάρχουν και ένα άλλο θέμα. Το ένα θέμα είναι το ζεστήρα σε ΣΥΝΑΠ που στόχο έχει να αποτρέψει την κρίση. Θα διαπιστώσετε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ήταν ο ίδιος. Το ΣΥΝΑΠ έχει μπει στην άκρη ενδεχομένως γιατί αφορά τις αγορές που προτιμάται που χρησιμοποιείτε. Εάν ε, μιλήσετε όμως και σε άλλους τομείς υπάρχουν θα σας πούνε ότι συμφωνούν με το ΣΥΝΑΠ γιατί τους δίνει ελαστικότητα μας λέμε ότι θα πρέπει να προστατευτούν από τον εαυτό τους. Το θέμα είναι τα ράνσεις και πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά. όπως βεστήρας είναι πάρα πολύ μεγάλος ή αν τον δεχτούμε στην πραγματικότητα απομακρύνουμε πολλούς ανθρώπους από την αγορά ΣΥΝΑΠ με εξαίρεση ορισμένους Αμερικανούς. Αμερικανούς. Θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στις Αμερικανικές τράπεζες. Από ό,τι φαίνεται το ΣΥΝΑΒ είναι ανασφαλές και το βίναθ είναι ασφαλές. Αλλά αν εξετάσετε τις έρευνες που αφορούν τις χρηματαγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένους ε, τομείς, στον τομέα της διάσωσης, θα έλεγα Εάν υπάρχει η εμπειρία της ε, διάσωσης, κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα τα δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Αν δούμε την εμπειρία των ΒΙΝΑΠΑ θα διαπιστώσατε ότι υπήρχε μια ε, διάσωση το 2007. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά αυτή την απλουστευμένη άποψη ότι το σύναφ είναι καλό, το βίναπ είναι κακό. Ιδιαίτερα όταν μιλάει κανείς στις εταιρείες, στις οργανώσεις που παρέχουν αυτά τα κονδύλια μιλάμε για μια λογιστική διαφορά. Το άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι θα συμβεί αν κλείσουμε το σύναβα. Πού θα, μετακινηθεί, θα μετακινηθούν αυτά τα χρήματα στο ΒΙΝΑΦ ή στο ε, τραπεζικό σύστημα. Ή θέλουμε να έχουμε μια συγκέντρωση του κινδύνου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διαφοροποιήσουμε το πού κατευθύνονται τα χρήματα ή να ε, μην συγκεντρώνεται σε επικίνδυνες ε, τράπεζες που όλοι μας γνωρίζουμε. Αν κοιτάξετε τους λογαριασμούς πολλών τραπεζών θα διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές δεν, ε, δεν είναι υγιείς και θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε περισσότερα κονδύλια σε αυτό το τομέα. Από την άλλη πλευρά έχω ορισμένες ανησυχίες ό,τι αφορά την αξιολογήσεις το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Όταν μιλάμε για CDO και για CDS, τα αποτελέσματα ήταν καλά και, πολύ, ε, και αυτό ενέπλεξε και πάρα, πολλού, πάρα πολλούς ε, ανθρώπους. Η αγορά όμως προηγήθηκε αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι αυτοί που χρησιμοποιούν και επενδύουν σε αυτούς τους τομείς έχουν τις δυνατότητες να κάνουν την αξιολόγηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα της ε, ρευτοποίησης και να σκεφτούμε και το θέμα των ε, ε, οίκων αξιολόγησης, στολυπτικής αξιολόγησης. <clears throat> Σας ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να παρέμβει για αυτό το θέμα. Εντάξει. Θα προσθέσω και εγώ τον εαυτό μου σύντομα στην παρέμβασή μου σε αυτόν τον κατάλογο αγοριτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε όταν ασχολούμεθα με αυτό το εγχείρημα ότι δεν θα έπρεπε, το είπε η Σιλβή, να δημιουργήσουμε ε, μια άλλη διαστρωμάτωση τραπεζών. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ποιο είναι. Είναι το ότι εξαρτώμαστε υπερβολικά από τις τράπεζες και δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση για τις αγορές αν είμαστε απρόσεκτοι στα όσα θα πράξουμε, αυτό το πρόβλημα θα επιδεινωθεί αντί να βελτιωθεί. Και συχνά λέμε κάτι ως προς το ότι ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες και κανονισμοί. Αλλά να θυμόμαστε ότι ο κίνδυνος εξαρτάται και από το ίδιο το θεσμικό όργανο στο οποίο εντάσσεται ένας θεσμός. Υπάρχει το ενδεχόμενο λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερο συστημικός κίνδυνος αν υπάρχουν μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες από ότι για παράδειγμα σε κάποια ταμεία που στο τέλος τέλος δεν θα κλειδονίσουν τις αγορές αν κάτι πάει στραβά όπως οι μεγάλες συστημικές τράπεζες. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, μπόρεσε να ανακάμψει από τη χρηματοοικονομική κρίση η αγορά της είπα, ταχύτερα από ότι σε εμά, για παράδειγμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας αναφέρουν ότι έχουμε συστημικό κίνδυνο στην Ευρώπη, μια και δεν έχουμε αρκετά ε, δραστηριοποιημένες με ενεργό χαρακτήρα αγορές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν να μην επιδεινωθούν τα πράγματα στην Ευρώπη από αυτούς τους συστημικούς κινδύνους. Να μην δηλαδή ε, κάνουμε κάτι το οποίο θα πάει στραβά. Έγιναν σχόλια τα οποία ανταποκρίνονται στη δική μου παρατήρηση. Θες να λάβεις τον λόγο εσύ λοιπόν τώρα σύντομα για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους σε αυτόν τον πρώτο γύρο ανταλλαγών απόψεων σε διμερές επίπεδο πρώτα και θα συνεχίσω φυσικά να ασχολούμαι και με αυτά τα θέματα σε σχέση με τους σκιώδεις εισηγητές ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο έκθεσης πολύ γρήγορα και θα μπορέσουμε να το διανύμουμε όταν θα έχουμε φτάσει εκεί και θα έχει οριμάσει. Θα επανέλθω και σε διμερείς επαφές που θα έχω για κάποια από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έγιναν σήμερα. Αλλά γενικότερα υπό τους όρους των παρατηρήσεων συμφωνώ πρέπει να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα είδους βάση, θεμέλια για να προχωρήσουμε και σε σχέση και με την ε, αξιολόγηση ή βαθμολόγηση και το πιο θεμελιώδες, θέμα φυσικά είναι το να υποστηρίξουμε περισσότερο την βίναφη, την σύναφη ή να μπορέσει να γίνει, να, γίνει πιο ε, δυσχερές στο πλαίσιο της σύναφ. Αυτά όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Και από πλευρά του συναδέλφου αναφέρθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο πορευόμαστε προς την, στο έργο αυτό που έχουμε αποδηθεί σε αυτό, κάποιες μελέτες ε, δείχνουν ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τους κινδύνους, την έκθεση στους κινδύνους και σε σχέση με τους, ε, τις ρυθμιστικές αρχές είναι σαφώς υπέρ της ΒΙΝΑΦ σε σχέση με το ΣΥΝΑΦ. Θα ήθελα να, θα να πάψει να λειτουργεί το ΣΥΝΑΦ όσον αφορά αυτού του είδους τους κινδύνους. Και συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται άμεση απάντηση στο ζήτημα τι θα γίνει αν τα ΣΥΝΑΦ δεν θα υπήρχαν πλέον, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λειτουργούν, τι θα κάναμε θα είναι ε, λιγότερο δημοφιλής αυτή η δραστηριότητα και θα, τα χρήματα θα πάνε τελικά αλλού ή υπάρχουν, ε, είναι αυτό περισσότερο επικίνδυνο. Τι θα γίνει. Είναι κάτι που και αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα σε υστερότερη φάση. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα έλεγα ότι το χρονοπλαίσιο έχει ήδη εξεταστεί και το έχουμε συζητήσει και στη συνέχεια με την, ε, το σχέδιο έκθεσης ε, θα το δούμε στις 2 Δεκεμβρίου και θα, στις 10 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα θα εκπνεύσει η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και έτσι τώρα καταφέρνουμε να προχωρήσουμε πιο μπρος ε, τα benchmarks δεν θα τα έχουμε παρά υστερότερα. Έχουμε χάσει κάποιους σκιώδεις εισηγητές. Δεν είμαι καν βέβαια ποιος είναι ο σκιώδης εισηγητή εισηγητής από τους Δεν το γνωρίζουμε ε, ποιος είναι. Προσπαθώ να το βρω και να δούμε αν κάποιος καλύπτει τη, από πλευράς του ΕΛΚΑ αυτό το έργο. Γκέι Μίτσελ λοιπόν, βρίσκεται καθοδόν ο Γκέι Μίτσελ θα έλεγα να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι ότου θα έχουμε την ευκαιρία να έχουν προσέλθει εδώ κάποιοι παραπάνω από αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Στις 4.30 λοιπόν θα ξαναξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε. Καθώς περιμένουμε έναν από τους χιώδεις εισηγητές, περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, δείκτες ως σημείο αναφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις. Είμαι σίγουρος ότι εδώ υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η έκθεση είναι δική μου. Σε κάθε περίπτωση Αφού είμαι συγγήτρια, καταρχάς θα ήθελα να πω ορισμένα πρακτικά θέματα. Καταβάλουμε μία προσπάθεια να καταφέρουμε κάτι τα κατά τη διάρκεια της θητείας, κάτι που ελπίζουμε όλοι και αυτό για να το πετύχουμε, συνέταξη το Σαββατοκύριακο το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών και τα έβαλα σε ένα έγγραφο, στο έγγραφο της, το της Επιτροπής ε, που ήδη έχει κυκλοφορήσει στους ε, σκιώδες. Όσοι λοιπόν θέλουν μπορούν να του δείξουν μια ματιά μετά από αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων. Αύριο θα το βάλω στην ιστοσελίδα μου έτσι ώστε όλοι να μπορούν να το πάρουν. Ε, εγώ δεν μπορώ να δώσω πολλές συνεδριάσεις, αλλά οι απόψεις που υιοθετώ θα είναι απόλυτα σαφείς και βεβαίως τα σχόλια θα γίνουν δεκτά. Πόσες επιπρόσθετες αραγές θα μπορούσα να δεκτώ πριν να υποβάλω την έκθεσή μου. Είναι κάτι που δεν ξέρω. Ενδεχομένω ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος, αλλά υπάρχει ένας γύρος τροπολογιών και ελπίζω ότι θα μπορώ να αρχίσω να δέχομαι μερικές που προέρχονται από άλλα ε, σημεία. Και βεβαίως θα τα δημοσιεύσω και στην ιστοσελίδα και θα δημοσιευτούν και άλλα έγγραφα έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν άποψη γι' αυτά. Βεβαίως θα καταλάβετε ότι έχω βασικά προωθήσει τις ε, δικές μου αρχές, τη δική μου προσέγγιση και θα σας πούμε λίγα λόγια τι έκανα. Το πρώτο πράγμα που έκανα αφορά το, το πεδίο εφαρμογής και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε πάρα πολλά ε, θέματα ενώ δεν έδωσε τον απαιτούμενο αριθμό δικτών αναφοράς Πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με έργα σε εξέλιξη. Αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να επικεντρωθώ στους διαχειριστές και στο άρθρο 5 όρισα μία σειρά από κατηγορίες δικτών αναφοράς αν ε, ο δείκτης αναφοράς πληρεί ένα από αυτά τα κριτήρια, τότε σημαίνει ότι εντάσσεται στον κανονισμό. Υπάρχει ένας κατάλογος στην αρχή του άρθρου 5, συμπεριλαμβάνει βεβαίως ε, σημαντικούς δείκτες, για την ώρα συμπεριλαμβάνει αυτούς των βασικών αγαθών. Είναι ευρύτατος και θα πρέπει να τον περιορίσουμε. Οι ιδέες βεβαίως είναι ευπρόσδεκτες. Αν ε, υπάρχει κάποια βασικός δείκτης αναφοράς και κατά την άποψή μου βασικός δείκτης αναφοράς είναι αυτός που ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια. Ένας αριθμός ε, που τον εφήβρα. Δεν ε, συμπεριέλαβα, δεν ε, υπολόγισα πόσους δείκτες ανεφορά συμπεριλαμβάνει. Ενδεχομένως θα μπορεί να έχει κανείς περισσότερους δείκτες. Σε κάθε περίπτωση συμπεριέλαβα ορισμένους για να μπορέσετε να ρίξετε μία ματιά γιατί κανένας ε, άλλος δεν βρήκε κάποια διαχωριστική γραμμή. Ενδεχομένως θα πρέπει να κινηθούμε προς τα ψηλά και όχι προς τα χαμηλά. Γιατί ένα από τα άλλα κριτήρια που έχω είναι ότι οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να πούν εγώ θα ήθελα να εντάξω αυτό μέσα στον κανονισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και μετά να επιταχύνουμε. Επίσης, έχω βάλει διαχειριστή που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα χρησιμοποιούνται στι αγορέ λιανικού εμπορίου. Αυτό είναι κάτι γενικό. Αν θέλουν να σκεφτούν, να σκεφτείτε πώ μπορούμε να το περιορίσουμε, βεβαίως και θα μπορούσα να το συζητήσω. Έχω αναφερθεί σε swaps και, άλλες συγκρίσιμους, και άλλους συγκρίσιμους δείκτες αναφοράς. Βεβαίως όλα αυτά είναι σημεία που θα πρέπει να αποδείξουμε. Έχω επίσης συμπεριλάβει διαχειριστές ε, δικτών που δεν έχουν ε, συναλλακτική φύση και <coughs> θα είναι ενδεχομένω ευεπηρέαστη ή δείκτες αγοράς που έχουν επίπτωση στην ενιαία αγορά. Ε, θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Θα ε, έλεγα ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε ορισμένες έννοιες, το να πούμε τι συμπεριλαμβάνεται εδώ και τι δεν συμπεριλαμβάνεται από τη στιγμή που ένας διαχειριστής συμπεριληφθεί στον κανονισμό, τότε ο κανονισμός ισχύει για όλους τους δείκτες αναφοράς. Ο λόγος που το προτείνω αυτό οφείλεται στο ότι αν παρέχει κανείς ένα σημαντικό δείκτη αναφοράς, έχει κάποια φήμη, κάποιο όνομα που θα χαρακτηρίζει όλους τους δείκτες, είτε είναι πάνω από αυτό κατόφλι ή όχι. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός. Θα μπορούσα λοιπόν να υπάρχουν κατευθυντήριοι γραμμές. Βεβαίως ε, το θέμα της αναλογικότητας εφαρμογής είναι θέμα ε, που θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Μετά η έγκριση στο άρθρο 23. Μόλις ξεπεράσει κανείς ε, αυτή την κατηγορία του δίκτυ αναφοράς. Αν θέλετε να εφαρμόσετε την αναλογικότητα, τότε ενημερώνετε την αρμόδια αρχή στο αίτημα έγκρισης ότι αυτοί είναι οι δείκτες αναφοράς και αυτό ακριβώς κάνω σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα και αν η αναλογικότητα να ζητηθεί και για τους άλλους που θα μπορούσε να είναι κάτι γενικό, τότε αυτό θα, θα υπάρχει μια εξήγηση για το πώς γίνεται η αρμόδια αρχή, θα μπορούσε να συμφωνήσει ή να μην συμφωνήσει. Προβλέπω ότι τις περισσότερες φορές θα υπάρξει μία συμφωνία. Και στο μέλλον, όταν θα γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε ορισμένα πράγματα, εάν ε, θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία δικτών στη ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε, έχω τη συνείδηση ότι επειδή είμαστε ε, ακόμα σε φάση πορεία και πολλές χώρε δεν έχουν νομοθεσία, θα υπάρξουν ε, διαδικασίες που θα πρέπει να περνάνε από τους ε, επόπτε και ότι ενδεχομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια ΙΟΣΚΟ. Η πρότασή μου είναι τα πρώτα πέντε χρόνια οι διαχειριστές να εξηγήσουν το πώς ε, θεωρούν τις, ε, ε, τους δίκτες αναφοράς και το πώς πληρούν τα κριτήρια της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων. Βεβαίως, υπάρχει ένας κατάλογος που έχει φτιάξει η ΕΣΜΑ και υπάρχει και μια πρόβληψη αντιστοιχίας. Αρχικά λοιπόν έχουμε ένα ανοιχτό πλαίσιο το οποίο βασίζεται στην Ιόσκο και οι αντιστοιχίες θα μπορούσαν να κινηθούν παράλληλα. Βεβαίως είναι κάτι που προσφέρεται σε, ε, ανοιχτό σε αμφισβήτηση, δηλαδή η υπόθεση που προέρχεται από την ε, ε, από αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσει. Στην πρόταση προ... λέμε στο διάστημα των 24 μηνών για την ε, υποβολή αιτήματο έγκρισης. Αυτό το πήρα σαν αρχική γραμμή για το benchmark για το δίκτυο αναφοράς ε, για τρίτες χώρες. Εδώ αναφέρομαι στους 30 μήνες. Η λογική μου είναι ότι πήρα αυτό που είναι στην τετράγωνη παρένθεση, 24 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι ότι χρειάζονται 3 μήνες για τη διαδικασία έγκριση και μετά προσέθεσα άλλους 3 ε, μήνες. Έτσι έφτασα στους ε, 30 μήνες. Βλέπετε ότι προσπαθώ να σας καταστήσω όλο πιο σα... όσο γίνεται πιο σαφή τον τρόπο σκέψης. Ένα-δύο πράγματα. Κώδικας διαοντολογίας, το άρθρο 9. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι ανάδεικτη αναφορά. Δεν είναι σαφές το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ή όχι. Ο κώδικας συμπεριφοράς από έναν διαχειριστή θα μπορούσε να γενικευτεί Και αν υπάρχει αναλογικότητα, τότε θα μπορούσαν να υπάρχουν ορισμένα σημεία που να μην είναι σχετικά. Προβληματισμοί σχετικά με το πώς θα υπάρξει νομική ε, δέσμευση. Ε, αυτό δεν γίνεται σε μία βάση... Προσπαθώ να πω ότι αυτό θα είναι όσο γίνεται πιο δεσμευτικό, αλλά θα πρέπει να είναι και πρακτικό. Θα πρέπει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να, οι διαχειριστές να γίνουν επόπτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Νομίζω ότι δεν είναι μια κατάλληλη δουλειά. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει κάποια γνώση, δηλαδή να μην λαμβάνονται μόνο πληροφορίες από ε, πηγές ε, που δεν έχουν υποβληθεί σε κάποιον έλεγχο. Αυτό θα πρέπει να αφορά την δέουσα επιμέλεια και θα πρέπει βεβαίως να τους απασχολήσει και το θέμα των υποβολών αυτών με ένα κατάλληλο τρόπο για να δουν αν υπάρχει κάτι λάθος στο μοντέλο και να αναφέρουν κάποια κατάχρηση, καταχρηστική συμπεριφορά στην αγορά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι δουλειά τους ε, να εξετάζουν τα πράγματα σε ένα πιο ε, ουσιαστικό επίπεδο. Στο άρθρο 12, στα παρατήματα, υπάρχει ένας τομέας που νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα τη συμμόρφωση προς τα κριτηρία της ΙΟΣΚΟ. Εγώ θα ήθελα να έχω την άποψη ε, αρκετή των ε, συναδέλφων αλλά και από τους stakeholders σχετικά με το πού θα μπορούσαν να ανακύψουν προβλήματα. Έχω ορισμένε ε, σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα την όλη αυτή η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τους ε, κρίσιμους δείκτες αναφοράς, τροποποίησα τον ορισμό για να τον καταστήσω πιο σαφή. Δεν άλλαξα αυτό το κατόφλι του 20% που λέει ότι αν χάσετε το 20% τότε υπάρχει μια υποχρεωτική διαδικασία. Με απασχολεί ότι αυτό το 20% ενδεχομένως είναι πάρα πολύ ψηλό ή πάρα πολύ χαμηλό. Εάν ε, ε, ε, υποθέτει κανείς ότι έχει εισρωές από όλη την Ευρώπη και χάσει μια γωνιά, έχει άλλη βαρύτητα. Εγώ θα έλεγα να το τροποποιήσουμε αυτό για να το γενικεύσουμε. Περιμένω. Λοιπόν, δεν το έχω τροποποιήσει όπως ε, είπα. Ε, το τι είναι δηλαδή ένα κρίση, ένας κρίσιμος δείκτης αναφοράς. Σε ό,τι αφορά μια δήλωση για το δίκτυο αναφοράς, το άρθρο 15, θα πρέπει να γνωρίζετε τι είναι οι δείκτες σας και να κάνετε κάποια δήλωση, ακόμα και όταν δεν πρόκειται για μεγάλους δείκτες. Δεν μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε κατά πόσον υπάρχει διακριτική ευχέρεια ή όχι. Το τροποποίησα αυτό, αν είναι κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί, ε, θα πρέπει να πούμε αν προσφέρεται ή δεν προσφέρεται ε, για έλεγχο. Στο άρθρο 39 βλέπω το... ότι το 50% δεν ε, είναι λειτουργικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι δείκτες αναφοράς θα πρέπει να ισχύσουν μέχρι την εκπνοή πολλών συμβάσεων. Ε, ενδεχομένω μιλάμε για 200 χρόνια και ενδεχομένω θα μπορούσε να προκύψει κάποια άλλη νομοθεσία. Για πρακτικούς λόγους θα μπορούσε κανείς ε, να περάσει αυτό το 5% και νομίζω ότι πολλοί θα αναρωτηθούν αν θα ανήκουν στο 5% όταν έχουν να κάνουν με μία σύμβαση. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να αφορά την καταγγελία. Λέμε τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά αυτά τα σημεία. Εγώ ε, αναφέρθηκα σε ορισμένα ορισμένε τεχνικέ προδιαγραφέ. Υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Ενδεχομένω όλοι δεν το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Είναι, ήταν η δικότητά μου πριν ε, γίνω Ευρωβουλευτή. Ε, δεν έχω κάνει τίποτα σημαντικό σχετικά με το θέμα αυτό. Ενδεχομένω δεν χρειάζεται κιόλα. Διευκρινίστηκα ότι ότι με βάση την αρχή της αποκάλυψης των δεδομένων δεν είναι αποκάλυψη της μεθοδολογίας και περιμένω να ακούσω τη δική σας άποψη για να διαπιστώσω εάν υπάρχουν ορισμένες άλλες ε, ε, προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν τίθεται θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα έλεγα όμως ότι θα πρέπει να γίνει κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών Λοιπόν, ε, θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο. Σε γενικέ γραμμές, αυτά έχω κάνει μέχρι τώρα, όπως σα έλεγα, μπορείτε να το βρείτε στο έγγραφο της Επιτροπής. Υπάρχουν και ένα-δυο άλλα πράγματα που θα μπορούσατε να δείτε, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι συνεκτικό και δεν χρειάζεται να γίνει κοινοποίηση συγκεκριμένων δικτών αναφοράς, γιατί όλα αυτά καλύπτονται από τη διαδικασία αδειοδότησης. Διαγράφεται συνεπώς το, το άρθρο 25. Ελπίζω να έχουν κάποιο νόημα αυτά που είπα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις συγητές. Ευχαριστώ Πρόεδρα για την λεπτομερέστατη εισαγωγή και για το σημείωμά σα ε, προηγουμένω που ήταν και τα δύο εξαιρετικά χρήσιμα. Βεβαίω και θα συνεργαστούμε μαζί σα για να καταλήξουμε σε ώστε να το πιο ικανοποιητικά συμπεράσματα σε αυτό το σύγχρονο χρονοδιάγραμμα που αναφέρατε. Ελπίζω να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Θέλω να θίξω κάποια ε, σχόλια εδώ. Πρώτον, να πω ότι είναι σαφές ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν ε, αμφισβητήσει, έχουν θέσει ένα αμφιβόλο την ακεραιότητα ε, των πιο σημαντικών των πιο σημαντικών τέτοιων δικτών ε, του Euro Interbank Rate και το καθεξής. Και αυτό οδήγησε σε απώλειες και εκατομμυρίων ε, δολαρίων και ευρώ και αντίστοιχα πρόστιμα. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το αναφέρουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αποκαταστήσουμε την ακεραιότητα του συστήματος. Και η έκθεση Άσκοτ αυτό το ανέφερε πολύ συγκεκριμένα για πάνω από 160 εκατομμύρια για μια εταιρεία, 59,5 εκατομμύρια δολάρια για άλλη και ούτω καθεξής. Πρέπει να το διευθετήσουμε λοιπόν. Πέραν του γενικού σημείου που πρέπει να εξετάσουμε που αφορά τους οίκους αξιολόγηση ε, και τι κάνουν. Πρέπει όμως πέραν τούτου να δούμε τι είδους κώδικα διοντολογίας αποκτήσαμε από τις ε, σχολές μας. Εκεί πρέπει να επιστρέψουμε. Να μην το αφήσουμε μόνο στην ε, ακαιρεότητα της αγοράς και τη χειραγώγηση της αγοράς που παρατηρήσαμε. Υπήρξαν ε, πολλές, ε, πολλά αιτήματα για συζητήσεις, για συναντήσεις, όμως όλες αυτές οι συναντήσεις αφορούν τον κλάδο, κυβερνητικούς φορείς, και το αναφέρω γιατί πρέπει να προσέξουμε. Γιατί κανείς δεν σκέφτεται τι θα γίνει με τους ε, δανειολήπτες, για παράδειγμα. Και τι είδους αντίκτυπο θα έχουν αυτές οι εξελίξεις στους δανειολήπτες. Δεν προτείνω να ε, τα βάλουμε όλα στο δύο καζάνι, ούτε θέλω να είμαι ιδιαίτερα επικριτικός, όμως πρέπει να βασιστούμε στη λογική για να δούμε πώς θα οριοθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Τούτου λεχθέντος η πρόταση της Επιτροπής γενικά συνάδει με τις αρχές ΑΙΑΣΚΟ για επέκταση ε, του πεδίου εφαρμογή να καλύπτεται μεγαλύτερη ποικιλία ε, benchmarks τέτοιων ε, φορέων αναφοράς. Οι αρχές, η ΆΣΚΟ προβλέπουν και ένα βαθμό ευελιξίας, γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, αποκλίνοντων των κανόνων που θα κατακαιρματίσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογή. Ίσως να μην συνάδουμε με τις κατευθυντήρες γραμμές ΕΣΜΑ για τα ETFs και άλλους χρήστες για τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται σε διεθνή φόρα όπως ο ΙΑΣΚΟ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διευκρίνηση τις επόμενες εβδομάδες πριν ε, ε, προχωρήσουμε στην εξέταση των τροπολογιών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο μπορεί να μην έχει εξετάσει η Επιτροπή, την εφαρμογή στα indices ε, στους δείκτες που παράγουν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. όπως ε, ο ε, δείκτης καταναλωτικών τιμών και ούτε καθεξής. Και αυτό μπορούν ε, να χαρακτηρίσουν τις επιδόσεις της εθνικής οικονομίας. Κατά τη φάση διαβουλεύσεων η Επιτροπή δεν ήθελε να συμπεριλάβει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Όταν δημοσιεύθηκε όμως ο κανονισμός δεν υπήρξε ρητή εξαίρεση για τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Όμως εφόσον επιβλέπονται από την Eurostat και ήδη υπάρχουν πολύ αυστηρά πρότυπα σε ό,τι τη μεθοδολογία και τη διαφάνεια, θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα κατά τη γνώμη μου. Γενικά, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι Ανησυχώ για το θέμα όσον αφορά τις διατάξεις για τους πληροφοριοδότες. Πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει αρκετά για τους πληροφοριοδότες. Και όσον αφορά τις αρχές για το benchmarking, τις βέλτιστες προδιαγραφές, από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Το έγγραφο προτείνει τα εξής θα πρέπει από πλευρά τη διοίκηση να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για τους πληροφοριοδότε, καθώς και διαδικασίες για παράπονα και προσφυγές ώστε να συνειδητοποιούμε νωρίς, ε, νωρίς το δυνατόν για τις παρατυπίε και τις, ε, τα οποιαδήποτε προβλήματα. Δεύτερον, ε, ο υπεύθυνο θα πρέπει να θεσπίζει ένα ποσοστό μηδενικής ανοχής, καθώς επίσης και πειθαρχικά μέτρα για τη μη συμμόρφωση, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική ε, πολιτική για πληροφοριοδότες. Και τρίτον, όσον αφορά ένα benchmark ε, υπολογισμό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ώστε να συνειδητοποιούμε αμέσως ε, τις οποιασδήποτε παρατυπίες και ανομαλίες μπορούν να ανακύψουν, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αποτελεσματικά. Η χειραγώγηση όσον αφορά στοιχεία από πλευράς ενδοπληροφόρησης προέρχονται από μια εφημερίδα την Guardian της Μεγάλης Βρετανίας με στοιχεία από πληροφοριοδότες. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ε, κινδύνους. για ένα καταστατικό για το πώς μπορούν τέτοιου είδους στοιχεία να αντιμετωπίζονται, πιστεύω ότι θα πρέπει με βάση τις αρχές ε, του benchmarking ε, να προχωρήσουμε ώστε να είμαστε κάπως πιο σοβαροί στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά τους ελέγχους, ε, καλοδεχούμενη είναι η πρόταση και οι προτάσεις που υποβάλλονται όσον αφορά την αναθεώρηση σε σε τακτική βάση και θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι η εξειδικευμένη αυτή δραστηριότητα θα είναι αποτελεσματική. Πρόεδρε, αυτά είναι τα γενικότερα σχόλια θα έλεγα που έχω να κάνω και που θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τα όσα εσείς τοποθετήσατε, θίξατε πιο πριν. Ίσως ένα θέμα τώρα που θα ήθελα να αναφέρω για τις απαιτήσει που ε, ζητούνται για την συμμόρφωση και κλεισμένων των θυρών ε, ε, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ε, αν αυτό θα έπρεπε να θυγεί τώρα και θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις και θα μπορούσα έτσι στη συνέχεια αν χρειαστεί να δώσω στους συναδέλφους τις παρατηρήσεις μου. Θα πρέπει να κινηθούμε το δυνατόν ταχύτερα. Τα θέματα τα οποία αναφέρατε είναι πράγματι θέματα θεμελιωμένα και πολύ θετικά. Και ελπίζω ότι από πλευράς θα ληφθούν υπόψη κάποιες από τις παρατηρήσεις που έκανα εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ε, έχετε εσείς τον λόγο Εμιλι. Ευχαριστώ Σάρον. Επίσης ε, και για το ανοιχτό πνεύμα και την προθυμία από πλευρά σου να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω από την ομάδα μας. Πρώτον όσον αφορά την ευρύτερη συγκυρία όσον αναφέρθηκε και από το ΕΛΚ προηγούμενα είδαμε τα σκάνδαλα από πέρυσι τα οποία ανέκυψαν. Τώρα έχουμε και την ε, περίπτωση όσον αφορά κάποιες απάτες, όσον αφορά συναλλαγές σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει ένα νομικό κενό εδώ που πρέπει να καλυφθεί οπωσδήποτε από πλευράς μας. Υποστηρίζουμε πραγματικά στεναρά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζονται αυτές, ε, ακόμα και μετά από πέντε χρόνια μετά από τη μεγαλύτερη κρίση έχουμε σε αυτό τον τομέα δυστυχώς πολλές απάτες ακόμα και χειραγώγηση περιπτώσεων με πολύ σοβαρό χαρακτήρα και αποβαίνουν εις βάρος των φορολογουμένων και θα πρέπει φυσικά να αντιμετωπίζονται. Και κάποια συγκεκριμένα πιο εξειδικευμένα σημεία σε σχέση με τα, το συνολικό ευρύτερο αυτό πλαίσιο, χειρώσεις για παράδειγμα η κυρία Αλήν Μακάτι έχει κάνει ήδη προηγούμενο έργο. Είναι πολύ σημαντικό τα επίπεδα κυρώσεων να μην ξεπερνούν αυτά τα οποία προτείνονται σε αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό. Πρέπει αυτό να είναι μια αρχή που θα μας εμπνέει και θα μας καθοδηγεί. Δεύτερον, υποστηρίζουμε όσο το δυνατόν ένα ευρύτερο πλαίσιο ένα ευρύτερο φάσμα και θα θέλαμε να εξετάσουμε φυσικά περαιτέρω τις προτάσεις σας όσον αφορά για την, τον περιορισμό αυτού του εύρου όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα πρέπει εξειδικευμένα σε βάθος να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Οι συνεχιζόμενες περιπτώσεις χειραγώγηση σε πολλούς τομείς ε, καταδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε ένα το δυνατόν ευρύτερο πλαίσιο όσο το δυνατόν ευρύτερο μπορεί να γίνει όσον αφορά τα διαφορετικά προϊόντα και τις πιο διαφορετικές αγορές αλλά πρέπει να τραβήξουμε και μια διαχωριστική γραμμή όσον αφορά το μέγεθος και θα εξετάσω φυσικά, θα εξετάσουμε τις προτάσεις σας. Είναι πολύ δύσκολο να τραβήξουμε μια ακριβή διαχωριστική γραμμή πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, για τα στοιχεία και τη μεθοδολογία που βρίσκονται στον τεχνικό πυρήνα αυτής της πρότασης, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα αυτό. Έχει κέρια σημασία, θεμελιακή σημασία αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα στοιχεία δεν έχουμε τίποτα στο χέρι μας. Αναφέρεται και κάποια στοιχεία επίσης όσον αφορά την αποκάλυψη, την δημοσιοποίηση στοιχείων και για την μεθοδολογική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετείτε γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε καταχρήσεις, καταχρηστικές περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να υπάρχουν τέτοια αιτήματα για την δημοσιοποίηση και στοιχείων και μεθοδολογίας στο σωστότερο επίπεδο ώστε οι αρμόδιοι να μπορούν να έχουν κάποιες δυνατότητες ε, να εξετάσουν αυτά τα θέματα και φυσικά και οι αρχές ως οι σημαντικότερα εμπλεκόμενοι για την προστασία των καταναλωτών. Εμείς ε, θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι η ενδεδειγμένη. Ε, εντάσσεται και στον κανονισμό MIFID. Εξετάζουμε να δούμε αν θα έπρεπε να ενταχθεί επίσης ε, και κάποια διάταξη ώστε να έχουν δικαιώματα αποζημιώσεων οι καταναλωτές όσον αφορά διατάξεις, κάτι το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν και από εθνικές οργανώσεις και συλλόγους και εξετάζουμε αυτή την πτυχή για την εποπτεία τώρα και για τις διαδικασίες αδειοδότησης όσον αφορά τις διοικητικές αρχές, τις αρμόδιες αρχές. Υποστηρίζουμε και υπήρξε και ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τον ρόλο του ΕΣΜΑ αν είναι αρκετό, αρκετά ισχυρό στη νέα πρόταση και για την προηγούμενη πρόταση ΛΙΚ που ήταν ισχυρότερη. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συμβιβασμός εντάξει βαίνει καλός αλλά πρέπει να έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο ενδυναμωμένο ρόλο για την ΕΣΜΑ ώστε να διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη εποπτεία όσον αφορά τις ε, πιο αποτελεσματικές διατάξεις και συνεργασία και με τις εθνικές αρχές ε, από πλευράς ε, ΕΣΜΑ θεωρούμε ότι είναι καλώ η πρόταση αυτή ως λύση αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο οι δυνατόν. Αυτές είναι οι γενικότερες ιδέες από πλευράς μας. Πρέπει γοργά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δούμε τις περαιτέρω λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Έφυγε, αποχώρησε ο Φιλίπ. Εσείς ε, θα τον αντικαταστήσετε, θα μιλήσετε εξ ονόματός του. Μόνο πολύ σύντομα θα μιλήσω εξ ονόματος του Φιλίπ και θα δώσω τις ακριβέστερες ή θα έχετε ακριβέστερο feedback στη συνέχεια. Λοιπόν, ξέρω τα γερμανικά δεν είναι ίσως η πιο όμορφη σε εισαγωγικά γλώσσα, τελκτική γλώσσα, σχολεία εκτός μικροφώνου. Ναι. Μην αρχίσουμε τώρα με τις, διαλο... με τις διαλέκτους του, της Ρινανίας Παλατινάτου. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι καλύτερο τώρα με τα γερμανικά ή όχι. Ε, okay. Μάλιστα, πολύ καλά. Λοιπόν, ο Φιλίπ σήμερα δεν μπορεί να παραστεί. Τα ακριβή σχόλιά του θα σας δοθούν στη συνέχεια γραπτός, ιστερότερα αλλά θα ήθελα δύο-τρία πράγματα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα θερμές ευχαριστίες για τον τρόπο που εργαζόμαστε και συνεχίζουμε το έργο έγκαιρα να μπορέσουν να ακουστούν αυτές οι παρατηρήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρόταση ότι και περαιτέρω δείκτες από τον τομέα των κεντρικών τραπεζών, των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών και των συστημάτων του συστήματος ευρωπαϊκών κεντρικών ε, τραπεζών εντάσσεται και μια μεγαλύτερη, ένας περισσότερο ανοιχτός χαρακτήρας ε, για τέτοιου είδους δείκτες και από ε, τρίτες ε, πηγές κεντρικών τραπεζιτών. Πρέπει με τέτοιου είδους δείκτες να μπορέσουμε να εργαστούμε και αναφέρθηκε αυτό πρόεδρε να δούμε ακριβώς τι σημαίνουν όλα αυτά τα 100 δισεκατομμύρια. Ποιος θα καλύπτεται και ποιος δεν θα καλύπτεται. Πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ εξειδικευμένα. Να μην χάσουμε κάποιον που πρέπει να συμμετάσχει που τελικά μπορεί να μην συμμετάσχει, να μην ενταχθεί. Και τι θα γίνει στο τέλος είναι περισσότερο τεχνικό θέμα για τις τιμές κατόφλια που πρέπει να λειτουργήσουν. Κάπως μας ενοχλούν οι προτάσεις ε, για το άρθρο 25 όπου εμείς την πρόταση που υποβλήθηκε την κατανοούμε ως εξής, ότι θέλετε να διαγραφεί η υποχρέωση ενημέρωσης όταν θα έχουμε θέματα νέων δικτών. Πιστεύουμε ότι είναι πιο σκόπιμο να έχουμε μια επισκόπηση πανευρωπαϊκά. Ποιοι είναι οι δείκτες εκείνες οι οποίοι παρισφρέουν στην αγορά ως νέοι δείκτες. Αυτό είναι η δική μας ερμηνεία όσον αφορά την διαγραφή του άρθρου 25. Στο τέλος θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο στο οποίο η κυρία Τούρνεν αναφέρθηκε είναι το θέμα του ρόλου της ΕΣΜΑ. Πριν από τη δημοσίευση αυτής της πρότασης υπήρξε ένα σχέδιο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το σχέδιο προβλεπόταν ότι για τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς δείκτες ε, θα είμαστε άμεσα, θα υπάρχει άμεση αρμοδιότητα. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμη ρύθμιση για μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Τέτοιοι δείκτες που είναι ειδικά ιδιαίτερα ισχυροί και ε, ε, επηρεάζουν ε, το, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΣΜΑ να είναι αρμόδια για αυτούς και να έχει κυρίαρχο ρόλο. Για τα θέματα Λίμπορ που είδαμε ότι ανεφύησαν και ακούμε διαμαρτυρίες και από τη Μεγάλη Βρετανία δεν θέλουμε κανένα τρόπο η ΕΣΜΑ λέει το Λίμπορ να εντάσσεται ως αρμοδιότητα για τα επιτόκια στο, στην ΕΣΜΑ. Στο τέλος τέλος ε, υπαναχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκατέλειψε κάποιες προτάσεις ε, ε, και όσον αφορά ίσως θέματα και του Euribor. Δεν πρέπει όμως εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο να δεχθούμε μια τέτοια πορεία. Έχουν μεγάλη σημασία για την μια ενιαία εσωτερική αγορά αυτοί οι δείκτες, για μια κοινή εποπτεία. Τουλάχιστον αυτή είναι η θέση, πρέπει να είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για αυτή τη συζήτηση αυτή τη συζήτηση πρέπει να την διεξαγάγουμε στην Ευρωβουλή. Είναι λυπηρό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπακούει κάποια κελεύσματα μελών του Συμβουλίου και υπαναχωρεί. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο μπορούμε να συζητήσουμε κάποια θέματα, αλλά θα ανέμενα από τους εισηγητές ένα πιο στεναρό ρόλο και απόψεις για την ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, now for the ECR side τώρα στη συνέχεια um, Ευχαριστώ πολύ. Ένα άλλο παράδειγμα της Επιτροπής που άλλα λέει και άλλα κάνει. Πάρα πολύ γραφειοκρατία σε αυτό τον κανονισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πραγματικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται οι κανονισμοί, αυξάνονται οι δείκτες αναφοράς και αν θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πραγματικό πρόβλημα και όχι σε μία αύξηση των δικτών αναφοράς. Με συγχωρείτε που θα πρέπει να το επαναλάβω, το θέμα της τραπεζικής κρίσης δεν μας έχει απασχολήσει οι τράπεζες ε, πτωχεύουν η μία μετά την άλλη και 5-6 χρόνια μετά από την αρχή της κρίσης δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτό και πολλά άλλα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει πληθωρισμός, ε, αυτό το δέχονται όλοι, και νομίζω ότι θα πρέπει να μας, βρει, να μας βρουν σύμφωνες αυτές οι κατευθυντήριοι γραμμές. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος. Ε, η κοινότητα δεν θέλει να ε, ε ρυθμίσει μόνο τα e αλλά όλα τα σημεία αναφοράς. Δηλαδή μια, ένας κανονισμός που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις ε, φωνές για διάσωση που βγάζουν οι τράπεζες ε, ή στις κατηγορίες για χειραγώγηση. Πώς θα μπορούσαμε να τα όλα αυτά. Οι μεμονωμένες οργανώσεις δεν έχουν ε, αντίρρηση στο να συμβάλλουν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα επιλύσουμε. Όπως είπε ο Σκιώδης, η συζητητής, η έκθεση της κυρίας Μακάρθη, είναι απόλυτα συνεκτική και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για τρίτες χώρες. Ζούμε σε ένα παγκοσμιο, παγκοσμιωμένο περιβάλλον. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να δεχτούμε ε, άλλους ε, να παρέμβουν σε αυτό το τομέα. Χαίρομαι που βλέπω τις αρχές προτάσεις της Σάρων να δείχνουν ότι κινούμεθα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι καταλαβαίνουμε τις λεπτομέρειες των ε, προτάσεών σου. Ας επικεντρωθούμε στις, στους συστημικούς δείκτες αναφοράς. Ας έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν αντικείμενο χειραγώγησης. Ας μην χρησιμοποιήσουμε την κρίση σαν ένα, μια δικαιολογία για να γίνουν επιπρόσθετος και άλλοι κανονισμοί. Ευχαριστώ. Να περάσουμε και σε άλλους ομιλητές. Η Σιλβί και δεν ξέρω και κάποιος άλλος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς παρεμβαίνουμε εδώ σε ένα τομέα όπου υπήρξαν απάτη αυτές υπήρξαν συμπεριφερές οι οποίες οδήγησαν σε δικαστικές διώξεις. Δεν θέλω να πω ότι υπήρξε υπερβολική ρύθμιση, κάπου ξεφύγαμε και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο Ευρωπαίος πολίτης κάτι περιμένει από μας. Δεύτερον, το θέμα που θα είναι πιο δύσκολο είναι ο καθορισμός του πεδίου. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην επισέλθουν στον τομέα αυτό ε, φορείς που δεν έχουν εξοικείωση με τους δείκτες αναφοράς από την άλλη πλευρά, να μην ξεφύγουν αυτοί που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πιστεύω ότι το θέμα του πεδίου εφαρμογή είναι το πιο δύσκολο σημείο. Εγώ με υπέρ το να δώσουμε εξουσίες στην Ίσμα. Γιατί, Γιατί όταν μία αρχή τοποθετεί ε, φορείς εποπτείας οτιδήποτε φορά την εσωτερική αγορά θα πρέπει να δοθεί σε μία αρχή που είναι αρμόδια για τον σύνολο των χωρών, δίχως να ε, ξεκινήσουν έρηδες. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας τομέας που θα πρέπει να διερευνήσουμε, ότι η Επιτροπή για δικούς της λόγους δεν το έχει κάνει. Αυτό θα συνάδει με αυτό που έκανε ε, το, ήδη το Κοινοβούλιο. Right. Thank you very much. Uh, Any other members wishing to speak? No, I think uh, Philip Todd from the Commission has been uh, waving at me, so I... Η εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, Γνέφη. Να του δώσουμε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την επισκόπηση των αρχικών σας ε, σκέψεων και περιμένουμε με ανυπομονησία την έκθεσή σας. Σας ευχαριστούμε επίσης για τα όσα είπατε ότι θέλετε να εργαστείτε ε, με ταχύς ρυθμούς και να διευκολύνετε ή δυνατόν μια γρήγορη συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό, αποτελεί προτεραιότητα για μας. Έχουμε δράσει ταχαίως και είμαστε από τις πρώτες ε, περιοχές στον κόσμο που έχουν εφαρμόσει τα πρότυπα ΙΑΣΚΟ. και σε άλλες περιοχές του κόσμου θέλουν να μας μιμηθούν. Ας αναφερθώ σε μερικές από τις παρατηρήσεις που έγιναν σήμερα το απόγευμα. Σε ό,τι αφορά το πεδίο, πράγματι έχουμε προτείνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, πρώτο και πρώτα απ' όλα για να ευθυγραμμιστούμε με την ΙΑΣΚΟ, που υιοθέτησε και επίσης ευρύ πεδίο στα πρότυπα που υιοθετηθήκαν πέρσι τον Ιούλιο. Ουσιαστικά, ε, οι δείκτες αναφοράς που έχουν τους ίδιους κινδύνους και έχουν ε, τα ίδια σημεία βαλωτότητας και για να μην υπάρξει κίνδυνος ε, κατάχρησης, αυτοί οι δείκτες λοιπόν θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. Αυτό είναι το σημείο κίνησής μας. Από την άλλη βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογική προσέγγιση και αυτό το επιτυγχάνουμε με το να έχουμε συγκεκριμένους ε, κανόνες για τα IBORs, έχουμε παραρτήματα για τους ε, δείκτες αναφοράς ε, αγαθών, για, τους, για το πετρέλαιο για παράδειγμα. Έχουμε ειδική διάταξη για τα benchmarks με δεδομένα που αντλούμε από ρυθμισμένες αγορές προς αυτές τις, αυτούς τους δείκτες αναφοράς. Έχουμε ε, ειδικές διατάξεις για τους ε, κρίσιμους ε, δείκτες αναφοράς, critical benchmarks, και εκεί προβλέπεται και σημαντικός ρόλος της ΕΣΜΑ. Και τέλος έχουμε διάταξη για τα, επίπεδα, για τα μέτρα επίπεδου 2, όπου μπορούμε να μετατρέψουμε τους κανόνες ανάλογα με τους δείκτες αναφοράς. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί ευρύ συγγνώμη, πεδίο εφαρμογής, αλλά αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα τις διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών benchmarks. Για τους πληροφοριοδότες whistleblowers. Ε, το σημειώνουμε, αλλά εφόσον ε, αυτό το θέμα έχει ήδη επιληθεί ε, στον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, εκεί υπάρχει ήδη διάταξη που προβλέπει την προστασία αυτών των πληροφοριοδοτών που καταγγέλουν ε, καταχρήσεις. Όταν δηλαδή υπάρχει υποψία κατάχρησης, αυτό μπορεί να ε, αναφερθεί στις αγορές. Το σημειώνουμε λοιπόν, όμως ε, η Επιτροπή Οίκων το έθιξε μέσω της εισηγήτριας. Σε ό,τι αφορά την ισορροπία για τους ε, κρίσιμου ε, δείκτες αναφοράς, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια καλή ισορροπία. Αναφέρεται ότι αφορά και άλλα κρατημέλη, αφορούν και άλλα κρατημέλη αυτά, αυτοί οι κρίσιμοι δείκτες αναφοράς και θα συμμετάσχουν και στις ε, συζητήσεις, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, αυτά τα τρίτα κρατημέλη. Τώρα, αν υπάρξουν διαφωνίες μέσα σε αυτό το σύνολο επιμελητών College of Supervisors. Βεβαίω τότε θα τα συζητήσουμε περαιτέρω. Όμω ε, με τα χαρά να συνεργαστούμε μαζί σα και με τα μέλη. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω εν συντομία σε κάποια από τα ζητήματα που έθιξαν οι συνάδελφοι για τον γκέι. Ναι, ε, κατανοώ αυτό που λες για τους δανειολήπτες ότι δεν μπορούν να υποβάλουν ε, θέσεις και εκθέσεις σε εμάς. Γι' αυτό και εγώ ανέφερα αυτό το ζήτημα ε, των ε, διαχειριστών και ότι μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα με τα κριτήρια. Και διατήρησα και το κριτήριο της καταλληλότητας όταν πρόκειται για ένα δίκτυ που αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα λιανικής. Όπως ανέφεραν οι πράσινοι, εγώ ε, διέγραψα την εξαίρεση της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να δείτε μόνο ό,τι διαγράφεται, αλλά και ό,τι αναφέρεται κάπου αλλού. Στο άρθρο 5 στο 5.1 κάτω-κάτω έχω αναφέρει ότι ο ΕΣΜΑ μπορεί να παράσει κατευθυντήριες γραμμές βάσει και σε αρχή της αναλογικότητας και ότι αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει και κατάλογο των εξαιρούμενων ε, τύπων ε, φορέων. Και αυτό που εννοούσα ουσιαστικά ήταν οι κεντρικές τράπεζες και στατιστικές υπηρεσίες. Όμως ε, οι γενικές εξαιρέσεις ε, ίσως είναι υπερβολικές, γιατί πολλά συμβαίνουν και με τις κεντρικές υπηρεσίες. Γιατί έχουμε πολλούς δείκτες που παράγονται και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον μία σύγκριση για το κατά πόσο ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι ακόμα ένα πλήγμα ενάντια της μυστικότητας ε, των κεντρικών τραπεζών, αν θέλετε. Όμως, όπου υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα, τότε μπορούν βεβαίως να εξαιρούνται. Και εγώ συμφωνώ ε, για το whistleblowing. Έχω συμπεριλάβει μια επιπρόσθετη ε, διατύπωση, κάπου το θυμάμαι το έβαλα και αυτό. μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες διατάξεις όπως και αλλού ε, στην, ε, στην οδηγία για την ε, κατάχρηση των αγορών και το καθεξής. Όμως αν δείτε και τα πρόσφατα, ε, τις πρόσφατες εξελίξεις, όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο supervised agencies, που τη χάνουν δηλαδή πτίας. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν θέλουμε να υπάρξει σύγκρουση εδώ. Καλό θα ήταν να το εφαρμόσουμε. Για την Έμιλη τώρα και όσους ανησυχούν για το πεδίο. Δεν θέλω να διαγράψω κάτι γιατί ε, θέλω κάτι πολύ ήπιο. Θα διαγράφω γιατί έχουμε κάτι το οποίο είναι ήδη αναλογικό, εξισορροπημένο και πρακτικά εφαρμόσιμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τις αρχές της ΑΙΟΣΚΟ. Ναι, πρέπει να έχουμε το κατάλληλο επίπεδο ε, δημοσιοποίησης προς, και κοινοποίησης προς τις αρχές, πράγματι, για να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι φορά το ρόλο της ΕΣΜΑ, που ανέφερε και η Σιλβή και ο Σφεν, ίσως υπάρχει ε, έδαφος ε, για περισσότερες αρμοδιότητες ε, ΕΣΜΑ, περισσότερες κατευθυντήρες γραμμές και RTS. Εφόσον η καταξιδότηση πράξη προς την Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευρύες και καλό θα ήταν να έχουν αυξημένο ρόλο της ΕΣΜΑ. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όπως ε, ό,τι συμβαίνει με τους οίκους αξιολόγηση με 500 ενδεχόμενου διαχειριστές. Και δεν ξέρω πόσους έχει η ΕΣΜΑ, κάτω από 80 νομίζω. 100? Δεν ε, Πρόκειται για μια εφάπαξ έγκριση ή αξιολόγηση. Πολλά γίνονται, είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Αν έχουμε τέτοιου είδους εποπτικούς μηχανισμούς που θέλει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με χιλιάδες υπαλλήλους, τότε καλά θα ήταν. Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο τώρα. Και θέλουμε ε, οι εθνικές αρμόδιες αρχές ε, εν ευθέτω χρόνο να μεριμνούν τους ώστε να υπάρχει δεσμευτική διαμεσολάβηση όταν είναι απαραίτητη η επίλυση κάποιων υποθέσεων. Και εγώ έχω συμπεριλάβει μερικά στοιχεία ακόμα αρμοδιοτήτων του ΕΣΜΑ. Και τέλος προς το Φίλιπ, ναι, η Άσκο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρύ πεδίο, όμως υπάρχει αναλογικότητα που δεν αφορά μόνο την κλιμάκωση, όπως είπες εσύ. Είπες ότι έχουμε αναλογικότητα με το να έχουμε επιπρόσθετα στοιχεία. Έξτρα εδώ, έξτρα εκεί για τους ε, δείκτες αναφοράς και ούτω καθεξής. Όμως ε, δεν υπάρχει ευρύ, μεγάλος όγκος πληροφοριών για το πώς μπορούμε να τα προσαρμόσουμε όλα αυτά. Και από ό,τι κατάλαβα από τι της πράξης δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι αλλιώ. Εμείς θα πρέπει να ενσωματώσουμε τον κατάλληλο βαθμό αναλογικότητας. Εγώ θέλω να το κρατήσω ανοιχτό. Ανεξάρτητα από το πώς καταλήγουμε σε ένα δείκτη, εάν δεν λειτουργούν, πάντα υπάρχει μια ευελιξία για να έχουμε κάτι επιπλέον. Αλλά αν κατακλείσουμε και τις αρμόδιες αρχές με πληροφορίες, με κοινοποιήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες δείκτε αναφοράς, τελικά δεν θα μα βγάλει πουθενά αυτή η προσέγγιση και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Τίποτα βεβαίω δεν μας εμποδίζει από το να έχουμε ε, και άλλους ε, δείκτες αναφοράς ε, στη συνέχεια. Όταν δούμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, ποιος ακολουθεί την προσέγγιση του ΑΙΟΣΚΟ, ποιος ε, έχει διοικητικέ εξουσίε και το καθεξής. Θα σα στείλω όμω ε, ένα αντίγραφο των όσων έχω κάνει τώρα. Όμω μην μένετε μόνο στα όσα διέγραψα. Το 25 μπορεί να διαγράφει γιατί η ουσία συμπεριλαμβάνεται κάπου αλλού. Όμω, τι νόημα έχει να έχουμε κοινοποιήσει για όλου αυτού του δείκτε αναφορά όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με όσους παράγουν τους δείκτε αναφοράς, να διασφαλίσουμε ότι το κάνουμε τον σωστό τρόπο. Ρυθμίζουμε τους οίκου αξιολόγηση, αλλά όχι τα όσα παράγουν ε, εν είδη αξιολογήσεων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κατά τη γνώμη μου. Η μεθοδολογία πρέπει να είναι σωστή, το σύστημα πρέπει να είναι σωστό, Αυτά τα φροντίζουμε, τα εξετάζουμε, αλλά δεν παρεμβαίνουμε για να τους πείσουμε να ξανακάνουν αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Λοιπόν, ε, είναι ένα προσχέδιο των θέσεών μου. Η επίσημη εκδοχή θα δημοσιοποιηθεί για πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 5 Δεκεμβρίου. Θα υπάρξει εξέταση. Εγώ θα την καταθέσω μέχρι τις 14 και προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό παίρνετε από τώρα κάποιες πληροφορίες για να μπορέσετε να τα σκεφτείτε μέχρι τότε. Η εξέταση τροπολογιών θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου για να έχουμε ψηφοφορία στις 30 Ιανουαρίου και να πάμε στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο. Αν έχετε κάτι ιδιαίτερα απτό ε, και για το Συμβούλιο. Ίσως ε, στους πρώτους μήνες της ελληνικής προεδρίας μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ελπίζουμε να γίνει αυτό. Ωραία, ας προχωρήσουμε τώρα λοιπόν. Α, αυτά ήταν, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Εποπτείας. Σας ευχαριστώ.